Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη αφορά στι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Κομισιόν με θέμα προσεχή παγκόσμια διάσκεψη για τι διεθνεί τηλεπικοινωνίε τη Διεθνού Ένωση Τηλεπικοινωνιών και ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του Κανονισμού Διεθνών Τηλεπικοινωνιών. Καλωσορίζω την Κυπριακή Προεδρία και δίνω μέσα το λόγο στον Υπουργό κύριο ε, Λουκά Λουκά εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, οι διεθνείς κανονισμοί τηλεπικοινωνιών αφορούν θέματα που σχετίζονται με διεθνείς και όχι με χώρες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές των κανονισμών που σχετίζονται άμεσα με το γεχτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιασδήποτε αλλαγέ στους κανονισμούς οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την παγκόσμια διάσκεψη wikid στον ντουμπάι δεν αντιβαίνουν με την ισχύουσα νομοθεσία στην ευρωπαϊκή ένωση. επιπρόσθετα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το wikid σε καμιά περίπτωση δεν θα περιορίσει την ευρωπαϊκή ένωση ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη του κοινοτικού κεκτημένου. Ω Προεδρία του Συμβουλίου βρίσκομαι σήμερα ενώπιό σα για να σα διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει πλήρω του δύο στόχου εν ώψη τη πιο πάνω παγκόσμια διάσκεψη. Την αποφυγή και εναντίωση σε οποιαδήποτε σύγκρουση με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαβεβαίωση ότι το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αναπτυχθεί όπως εμείς επιλέξουμε τα 27 κράτη μέλη τα οποία θα συμμετάσχουν και θα διαπραγματευτούν στο WICIT ω πλήρη μέλη θα μεταφέρουν και θα υπερασπιστούν αυτά τα δύο μηνύματα στα άλλα 163 κράτη μέλη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU η οποία διοργανώνει αυτή την παγκόσμια διάσκεψη. Τα 27 κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα του ukip αντανακλά τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και των υφιστάμενων υποχρεώσεων. όπως γνωρίζετε η προπαρασκευαστική διαδικασία για το ukip είναι αρκετά περίπλοκη. ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή ένωση είναι η ομάδα εργασίας της itu και η διάσκεψη των διοικήσεων ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και η ευρωπαϊκή επιτροπή έχουν συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν την προπαρασκευαστική διαδικασία και υπερασπίστηκαν εκεί την ίδια γραμμή. η ευρωπαϊκή επιτροπή θα συμμετάσχει επίσης στο wikid όχι ως πλήρες διαπραγματευτικό μέλος αλλά ως παρατηρητής. η πλήρη συμμετοχή επιτρέπεται μόνο για τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της itu σύμφωνα με τους κανόνες της itu. ωστόσο προκειμένου να επωφεληθούμε περισσότερο από τη συμμετοχή της Επιτροπής στο WICIT στην προσπάθεια προάσπισης ή ρύθμισης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουμε στο WICIT όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Επιτροπής να γίνει δεχτή ως παρατηρητής με συμβουλευτική ιδιότητα. Παρά το γεγονός ότι αυτό το καθεστώς δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί επί των προτάσεων θα τη επιτρέψει να ζητήσει τον λόγο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αφού ολοκληρωθούν οι παρεμβάσει των κρατών μελών τη itu προκειμένου να παρέχει χρήσιμε συμβουλέ ή πληροφορίε σε σημεία που σχετίζονται και ευθυγραμμίζονται με τη θέση τη ευρωπαϊκή ένωση. από την ανάληψη τη κυπριακή προεδρία συζητούμε την πρόταση τη επιτροπή η οποία επί τη ουσία υποστηρίχθηκε πλήρω από το συμβούλιο αποφυγή και εναντίωση σε οποιαδήποτε σύγκρουση με το κεκτημένο της ευρωπαϊκής ένωσης και διαβεβαίωση ότι το κεκτημένο της ευρωπαϊκής ένωσης θα μπορεί να αναπτυχθεί ως εμείς επιλέξουμε. η επιτροπή πρότεινε επίσης ότι η ευρωπαϊκή ένωση που θα εκπροσωπείται από την επιτροπή θα πρέπει να διαπραγματευτεί την αναθεώρηση των κανονισμών στον Ντουπάι σε αυτό το τελευταίο σημείο ωστόσο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κανόνες της itu δεν επιτρέπουν στην ευρωπαϊκή ένωση να συμμετάσχει στο WICIT ως πλήρες διαπραγματευτικό μέλος. είτε η επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής ή ως παρατηρητής με συμβουλευτική ιδιότητα οι κανόνες της itu δεν επιτρέπουν στους παρατηρητές να υποβάλουν προτάσεις ή να διαπραγματευτούν θέσεις η απόφαση να επιτρέψει στην επιτροπή να συμμετάσχει ω παρατηρητή με συμβουλευτική ιδιότητα θα ληφθεί κατά την πρώτη ημέρα από τον πρόεδρο του συνεδρίου στο ντουμπάι. επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξή το συμβούλιο αναγνωρίζει πλήρω το γεγονό ότι η επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τη θέση τη ένωση αλλά μόνο τα κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν τι προτάσει αυτοί είναι οι κανόνε τη itu και το συμβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει αυτού τους κανόνε. αυτό που έχει σημασία είναι ότι η επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι η θέση της ευρωπαϊκής ένωσης θα παρουσιαστεί στον Τουπάι σωστά με συνέπεια και έγκαιρα με βάση τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη των συνέδρων που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. επομένως καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να μεριμνήσουμε για τον αποτελεσματικό συντονισμό επιτούτου προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στις πολλές προτάσεις που μέλη της itu σκοπεύουν να καταθέσουν. η κυπριακή προεδρία ετοίμασε άτυπο έγγραφο πρακτικών διευθετήσεων το οποίο συζητήθηκε στο συμβούλιο για την καλύτερη συνεργασία και τον συντονισμό των ενεργειών των 27 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Προς αυτόν τον σκοπό, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου συνδιοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντηση με τους επικεφαλείς των εθνικών αντιπροσωπιών των κρατών μελών ή εκπροσώπους τους στον Τουπάι, κατά την οποία έγινε σε βάθος συζήτηση των θεμάτων πρακτικής συνεργασίας και συντονισμού ενεργειών για την καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συνέδριο. Ελπίζω ότι οι απαντήσεις μου προς την διαδικαστική διάσταση του WIKIT κάλυψαν επαρκώς τα ζητήματα που τέθηκαν στην προφορική ερώτηση από το αξιότιμο μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, κυρία Φερχάιεν. Ως προς την ουσία, όσον αφορά τη ρύθμιση του διαδικτύου και την χρέωση των παροχέων περιεχομένου στο διαδίκτυο αρκεί να πούμε ότι στο Wikit θα συμφωνήσουν ότι η itu θα πρέπει να ρυθμίζει το διαδίκτυο και ότι οι παροχεί τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να χρεώνουν του παροχεί περιεχομένου στο διαδίκτυο. τότε αυτό θα ήταν σε αντίθεση με τον κύριο στόχο της ευρωπαϊκής ένωσης για το wikid αφού τα αποτελέσματα δεν θα είναι συμβατά με το γεχτημένο της ευρωπαϊκής ένωσης και τώρα αλλά και στο μέλλον. οι κοινέ ευρωπαϊκέ θέσει αντικατοπτρίζονται στι ευρωπαϊκέ κοινέ εισηγήσει όπω θα κατατεθούν στο συνέδριο από την ΣΕΠΤ, οι οποίε λαμβάνουν υπόψη και συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με την παρατήρηση ότι όταν οι διεθνεί κανονισμοί τηλεπικοινωνιών εγκαθιδρύθηκαν το 1988, αυτό έγινε σε ένα περιβάλλον με παραδοσιακά δίκτυα στη βάση μισθωμένων συνδέσεων με άλλα λόγια ξεχωριστά δίκτυα για ξεχωριστέ υπηρεσίε. στι μέρε μα όλο και περισσότερο υπάρχει μια ενιαία υποδομή με βάση το πρωτόκολλο διαδικτύου για την παροχή όλων των υπηρεσιών είτε πρόκειται για φωνή βίντεο ή δεδομένα και σε μια μόνο συσκευή. επιπρόσθετα υπάρχει δραματική αύξηση στην κινητή τηλεφωνία καθώς επίσης και αυξανόμενη συμφόρηση στα δίκτυα ως αποτέλεσμα της αύξησης στην κίνηση δεδομένων και ειδικά δεδομένων βίντεο. όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν προκλήσεις στη δομή των σημερινών συστημάτων επικοινωνιών και στους κανόνες που διέπουν τα εν λόγω συστήματα τόσο στον ανεπτυγμένο καθώς και στον αναπτυσσόμενο κόσμο το συμβούλιο δεσμεύεται πλήρως να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η έκβαση του wikid να είναι πλήρως σύμφωνη με το κεκτημένο της ευρωπαϊκής ένωσης και με το στόχο της ευρωπαϊκής ένωσης για την περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής οικονομίας στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ τον ε, εκπρόσωπο της προεδρίας τον εκπρόσωπο του συμβουλίου. Ε, το λόγο έχει ο επιτρόπος κ. αντώνιο ταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αντικαθιστώ σήμερα την Αντιπρόεδρο Νέλη Κρούς. Το διαδίκτυο που γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε σήμερα αναπτύχθηκε ε, χάρη στο στη δυνατότητα που δώσαμε στα δημιουργικά ταλέντα να χρησιμοποιήσει τις υποδομές προς όφελος ε, των πολιτών με Open Access. Επίσης είναι πηγή το διαδίκτυο οικονομικής ανάπτυξης ε, για πολλές ε, χώρες στον κόσμο και πολλές αναπτυσσόμενες. Στην προσεχή παγκόσμια διάσκεψη διεθνών τηλεπικοινωνίας του Ντουμπάι, μία, ίσως ε, θεσπιστεί μια πιο δεσμευτική ε, ρύθμιση για το ίντερνετ. Κάτι τέτοιο όμως ε, θα παραβλάψει την καινοτομία και την ανάπτυξη σε ένα τομέα που συμβάλλει πολύ στην παγκόσμια οικονομία και ίσως περιορίσει την ε, κυκλοφορία των δεδομένων και αυξήσει το κόστος, δημιουργήσει διοικητικά εμπόδια και περιορίσει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δεν είναι προς όφελός μας να καταπνίξουμε το τεράστιο κεφάλαιο που αποτελεί το ίντερνετ πολλές χώρες που θέλουν μεγαλύτερη ρύθμιση του ίντερνετ μέσω της διαδικασίας του Ντουμπάι δεν εστερνίζονται τις δικές μας αρχές και αξίες ε, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να ανοίξουμε στις χώρες αυτές το δρόμο για έναν αυστηρότερο έλεγχο του διαδικτύου ίσως δημιουργήσει κίνδυνο προσβολής της ελευθερίας έκφρασης, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της εύλογης έκφρασης και της πολιτικής, των πολιτικών αντιρρήσεων μερικές φορές. Για όλους αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εναντιωθεί σε μια διεύρυνση των ρυθμίσεων, ε, των κανονισμών για, την παγκόσμια, για τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της κυκλοφορίας των δεδομένων. Μάλιστα, συμμετείχαμε ενεργά στις προπαρασκευαστικές εργασίες της παγκόσμιας διάσκεψης, ε, της WICET, και περιμένουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις στο Ντουμπάι, εξαιτία των θέσεων πολλών χωρών και των προσδοκιών τους για μια νέα συνθήκη. Πολλές μάλιστα βέβαια χώρες ε, συμμερίζονται τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι αισιόδοξο ότι ε, υπερβολικά περιοριστικές ρυθμίσεις τελικά θα αποφευθούν. Χρειαζόμαστε επαγρύπνηση, ε, καλύτερο συντονισμό και φυσικά εργόδεις προσπάθειες μεταξύ μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται που η ΕΤΝΟ, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Παρόχων Τηλεπικοινωνιών και Ελεκτρονικών επικοινωνιών προσχώρησε στη θέση της ε, Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ταχυδρομικών Διοικήσεων και Τηλεπικοινωνιών που προβλέπει ότι τέτοιου είδους διατάξεις δεν έχουν θέση στους κανονισμούς για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια απόφαση του Συμβουλίου ε, για μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εν ώψη της ε, WICIT, της Παγκόσμιας Διάσκεψης Διεθνών Τηλεπικοινωνιών, υιοθετήθηκε στις 2 Αυγούστου του 2012 και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η θέση μας μεριμνά στο οποιαδήποτε αλλαγή του κανονισμού για τις, για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες δεν θα επηρεάσει τους κοινούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα τροποποιήσει την εμβέλειά τους και το πεδίο εφαρμογή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη πλατφόρμα το Wicked για να ε, καθοριστούν τα συστήματα τιμολόγησης ε, και ε, αποζημίωση αντισταθμιστικών μέτρων. Συγκεκριμένες διατάξεις για τις τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ουδετερότητα και την αμεροληψία του ίντερνετ που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητες. Τα κράτη-μέλη εντός ολίγου θα υιοθετήσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή αυτής της πρότασης που υπέβαλε η Προεδρία. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κρατημέλη εξέφρασαν ήδη την υποστήριξή του προ τη θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τέτοιε πρωτοβουλίε θα αποβούν ει βάρο τη μελλοντική ε, ανάπτυξη του Ιντερνετ, που είναι ανοιχτή πλατφόρμα και καινοτόμα πλατφόρμα επικοινωνία. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τη θλίψη τη για το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνίε για θεσμικά ζητήματα, όπω το θέμα της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Μια ισχυρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα χειρό μήνυμα θα είναι σημαντική ε, στο Ντουμπάι. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αφιστεί προσπαθειών προκειμένου να προασπίσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με στεναρό τρόπο ε, στην παγκόσμια διάσκεψη διεθνών τηλεπικοινωνιών στο Ντουμπάι. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Υμνάμεντε ΕΦΑΟΠΕ. Εξ ονόματο τη ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, το λόγο τώρα έχει η κυρία ε, συνάδελφο Σαμπίν Φερχάιν για δύο λεπτά. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο θα λάβει η χώρα η ε, Παγκόσμια Διάσκεψη για τι διεθνεί τηλεπικοινωνίε και θα αναπτύξει, θα συζητήσει νέε προδιαγραφέ. Μέχρι τώρα η ITU ε, είχε τις αρμοδιότητες. Ορισμένες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, κάποιες αραβικές ε, και ε, άλλες θέλουν ε, να μετατεθούν οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες και να ενταχθεί και το διαδίκτυο σε αυτές. Εμείς με το ψήφισμά μας θέλουμε να διατρανώσουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι για την ελευθερία της γνώμης, για την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των ιδεών ε, ε, θα πρέπει να ε, διαφυλάσσουν την ελεύθερη πρόσβαση και δωρεάν πρόσβαση. Πολλές φορές αυτό είναι μεγάλη αξία για την ανάπτυξη, για την ελευθερία της γνώσης, για την ανταλλαγή ιδεών και για την οικονομική δραστηριότητα. Έγινε πλέον το διαδίκτυο απόσπαστο τμήμα δημοκρατικών δομών. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν αγορές από το διαδίκτυο. Γι' αυτό καλούμε Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη WIKIT να μην διευρύνουν ε, τις ε, ε, αρμοδιότητες της ITU να καλύπτει και τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Θα πρέπει να γίνεται σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αισθητός και η δυνατότητα να αναπτύσσεται στο μέλλον το διαδίκτυο. Η διακυβέρνηση του διαδικτύου έχει εφαρμοστεί και αποδειχθεί στην πράξη επιτυχής μέσα από διάφορους φορείς, η λεγόμενη multi multi-governor, ε, Θα πρέπει να αναπτυχθεί η κοινοτική θέση και να παρουσιαστεί προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Ε, ακολουθεί στο βήμα εξ ονόματος της ομάδος S&D ο συνάδελφος κύριος Κάλφιν για δύο λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο Κοινοβούλιο αποτρέψαμε πριν από λίγο καιρό την έγκριση της άκτα και ψηφίσαμε με συνέπεια για την ελευθερία και το ανοιχτό ίντερνετ. Η επικείμενη Wiki, η Παγκόσμια Διάσκεψη Διεθνών Τηλεπικοινωνιών ε, του Δεκεμβρίου, ε, θα πρέπει ε, να μας βρει ενωμένους με ένα πολύ χειρό μήνυμα με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια ε, της ITU, που είναι ένα σώμα των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε πολλές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα που συμμετέχουν στην ITU. Σήμερα το διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο και πολλές χώρες ε, θα ήθελαν να το ελέγξουν επειδή φοβούνται πώς θα χρησιμοποιηθεί και θέλουν να περιορίσουν την ελευθερία των ανθρώπων να το χρησιμοποιούν. Έχουμε πολλές χώρες και οργανώσεις που θέλουν ε, να θεσπιστούν έλεγχοι για το διαδίκτυο, αλλάζοντας το επιχειρησιακό μοντέλο, καθιστώντας το πιο δαπανηρό και λιγότερο προσιτό και φυσικά ε, αυξάνοντας τα μονοπόλια σε αυτό. Ακούσαμε πριν από λίγο καιρό ότι κάποιε κυβερνήσει θέλουν να δημιουργήσουν εθνικό Ιντερνετ. Αυτό όμω είναι σχήμα οξύμορο, ε, ανέφικτο εξορισμού υποβληθούν πάντως από τη Ρωσία ένα πολύ ισχυρό κράτος σχετικές προτάσεις ε, στο Wikit και θεωρεί ότι οι κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν κυρίαρχα δικαιώματα να ελέγχουν τι υπηρεσίε που παρέχονται από το Ιντερνετ. Αυτό θα, θα δώσει ένα τέρμα στην ελευθερία του Ιντερνετ και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν, να διαχειρίζονται, να διακυβερνούν το Ιντερνετ στην εθνική του επικράτεια. Μα τι σημαίνει αυτό. Πώ θα μπορούμε να συνδέσουμε το διαδίκτυο με τα κυρίαρχα δικαιώματα μια χώρα. Επίση, υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την απόφαση ε, για τις ε, ε, διευθύνσεις και τα domain names στο ίντερνετ. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Επιμένουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά με μεγάλη συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο έχει συνάδελφος κυρία Σάκε για δυόμιση λεπτά. Technology. Thank ε, τεχνολογία που λέγαμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε για κανόνες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ουσία ε, για την κεντρική ιδέα του ψηφίσματος. Έχουν αλλάξει το διαδίκτυο και η τεχνολογία του τη ζωή των ανθρώπων παντού στον κόσμο. Ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες, ελεύθερη έκφραση ε, και καταγγελία ε, παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για επιχειρήσεις. Είναι πολύ συναρπαστικές οι δυνατότητες. μπορούν πιο εύκολα να προσβληθούν τα μονοπόλια και εξουσίες ε, των κυβερνήσεων ε, ε, πάνω στον τύπο. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργηθούν τώρα νέα μονοπόλια. Οι επαναστατικές αλλαγέ ποτέ δεν έρχονται χωρίς διαμαρτυρίες εκείνων που έχουν συμφέροντα. Και οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξασφαλίσουν το κερδοφόρο μοντέλο, αλλά και οι κυβερνήσει που θέλουν να ελέγχουν του λαού. Οι πολιεθνικέ και οι διεθνεί οργανισμοί είναι ο νέο στίβο για αυτέ τι μάχε. Ε, είναι μια τεχνική κάπως σκοτεινή ε, οργάνωση αυτή του ΟΗΕ που ασχολείται, αλλά είναι το θέμα πολιτική μάχη και επανατοποθέτηση του διαδικτύου που θέλουν να βάλουν χέρι τα κράτη-μέλη για να ελέγχουν τα μοντέλα τους ή να προστατεύουν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Και στο όνομα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί η παρακολούθηση ε, των πολιτών και περιορίζεται η ελευθερία της άποψης όταν ποινικοποιείται όπως είναι σε χώρες όπως είναι οι αφρικανικές χώρες ή ακόμα και στη δική μου χώρα την Ολλανδία παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Η διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ορισμένοι λέγουν ότι αυτό είναι μια αντίφαση και μόνο ως έκφραση. Δεν χρειάζεται το διαδίκτυο πολύ μεγάλη ρύθμιση. Ε, σήμερα συζητούμε πραγματικά ε, για την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών που συγκάλεσε τη διάσκεψη στο Ντουμπάι για την, ε, τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες και θα πρέπει βεβαίω να ενημερωθεί λίγο ο κανονισμός που ισχύει γιατί δεν έχει γίνει ενημέρωση εδώ και καιρό. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συστάσεις του ITU δεν είναι δεσμευτικά κείμενα. Προωθούν βέλτιστες πρακτικές. Τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν ε, μία ψήφο το καθένα και αν θέλει η Ένωση να είναι πραγματικά ενωμένη και να κάνει τη φωνή της να ακουστεί, θα πρέπει να ομονοήσουμε να είμαστε ε, σύμφωνοι και να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκε. Στον όνομα της ομάδας των Πρασίνων το λόγο έχει συνάδελφος κυρία Άντερς Ντότα για ένα λεπτό. Thank you, Chairman. Colleagues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να συζητήσει το θέμα της ε, επερχόμενης ε, διάσκεψης για τις διεθνείς επικοινωνίες. Το πώς θα πρέπει να επικοινωνούμε θα λαμβάνονται ως απόφαση το, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, δυστυχώς όμως ε, ξεφεύγουν από, τους, από το ευρύ και δεν τη χάνουν τις δέουσες προσοχής. Την ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του, ε, των πολιτών όσον αφορά τα ε, θέματα τηλεπικοινωνιών. Έχουμε ετοιμάσει και κάτι που αφορά τις ε, τεχνολογίες ε, του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών. Ασχολούμαστε και με το θέμα της διαφάνειας ε, στις διαδικασίες ITU και WIKID που αναφέρθηκε από το Συμβούλιο προλίγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των πολιτικών ομάδων για τη συνεργασία τους και ελπίζω το Συμβούλιο και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη τα σχόλιά μας στις μελλοντικέ τους εργασίες. Uh, Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκίναρ Χέκμαρκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το σημαντικότερο μας καθήκον είναι να προσπίσουμε την ελευθερία στο διαδίκτυο. Και Χαίρομαι ιδιαίτερω για την ομοφωνία που υπάρχει ως προς αυτό. Είπαμε όλοι ότι η ελευθερία στο διαδίκτυο είναι προϋπόθεση για την ίδια την ανάπτυξη, την περαιτέρω ανέλυξη του ίντερνετ. Και ε, ελευθερία του ίντερνετ σημαίνει ελευθερία στην κυκλοφορία των πληροφοριών, ελευθερία έκφρασης και αυτή η ελευθερία έχει αλλάξει και αλλάζει, αλλά θα αλλάξει και στο μόλιν της κοινωνίας μας. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να προασπίσουμε και να διαφυλάξουμε αυτή την ελευθερία του ίντερνετ. Υπάρχουν όμως πολλές δυνάμεις, πολλά καθεστώτα προσπαθούν να παρεμποδίσουν την εξέλιξη του ίντερνετ για τους λόγους που επισημάναμε, επειδή ακριβώς φοβούνται αυτή την ελευθερία έκφρασης που εξασφαλίζει το διαδίκτυο. Φοβούνται αυτή την ελεύθερη ροή πληροφοριών. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε σαφείς, κατηγορηματικοί και αποφασισμένοι να προσπίσουμε την ελευθερία στο διαδίκτυο. Επίσης, δεν θα πρέπει να δώσουμε προσχήματα και άλλοθε σε αυτούς που επιδιώκουν τις παρεμβάσεις στο ίντερνετ και τον περιορισμό της ελευθερίας. Θα πρέπει εμείς να μην έχουμε την ευκαιρία για να μπλοκάρουμε υπηρεσίες ή να δεχόμαστε κάτι που γίνεται αλλού. Γιατί έτσι κάτι τέτοιο θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα από τις δυνάμεις και τα καθεστώτα που ενδιαφέρονται να παρεμποδίσουν την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία πληροφόρησης και μπλοκάρουν την ίδια τη σημασία του ίντερνετ. Θα δούμε τις ίδιες αλλαγές στο μέλλον με αυτές που είχαμε και στο παρελθόν. Και ο καλύτερος τρόπος για να διαφυλάξουμε αυτή την ελευθερία είναι να την προασπίσουμε απέναντι σε οποιοδήποτε καθεστώς που θέλει να αναχαιτήσει την ανάπτυξη του ίντερνετ. Και χαίρομαι που έδειξαν αποφασιστικότητα και το Συμβουλίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Ακιάνη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, υπενθυμίσαμε το Δεκέμβριο ο Οργανισμός των Εθνών που ασχολείται με τις ε, τηλεπικοινωνίες ε, και το διαδίκτυο θα κάνει μια διάσκεψη στο Ντουμπάι για την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε και χαίρομαι ιδιαίτερα για τα όσα ακούσαμε από τον Επίτροπο Ταγιάννη, τα όσα αν έχουν γίνει μέχρι τούδε, τα οποία δεν θα πρέπει να αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση ούτε πρέπει να επιτρέψουμε οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, παρακαμφθούν από έναν ε, ε, διεθνή οργανισμό όπως είναι η ITU, στον οποίο γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν πολλά κράτη παγκοσμίω που όπως γνωρίζουμε έχουν προβλήματα με την ελευθερία έκφρασης και τη διαφάνεια. Είναι σωστό λοιπόν να λέμε ότι κινδυνεύουν οι πυλώνες ε, του διαδικτύου, η ελευθερία, η συμμετοχή, ο πολιτισμός και η κοινοτομία. Είναι απαραίτητο λοιπόν ε, να προστατεύσουμε το ρόλο του διαδικτύου και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το διαδίκτυο για την ανάκαμψη της ε, οικονομίας αλλά και για να διασφαλίσει και ίσες ευκαιρίε για όλου. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ως στόχο η Ευρώπη στο Ντουμπάι να, μιλεί, να μιλάμε μία ενιαία φωνή. Είναι πολλές οι αμφιλεγόμενες προτάσεις που παρουσιάζονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην ε, ε, Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνές Τηλεπικοινωνίες, ιδίω όσον αφορά τη διακυβέρνηση του διαδικτύου που αμφισβητούν την ιδιαιτερότητα του διαδικτύου με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές. Ο κίνδυνο λοιπόν είναι η ελευθερία του διαδικτύου ή πιο συγκεκριμένα η ελευθερία έκφρασης και προστασίας των δεδομένων. Αυτά τα οποία προτείνουν κάποια κράτη-μέλη επιτρέπουν ε, σε, στις κυβερνήσεις ε, να ε, όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στο πώς κάνουν χρήση στο διαδίκτυο. Έτσι ε, το χάσμα μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και λογοκρισίας είναι πάρα πολύ μικρό και γι' αυτό θα πρέπει να προσπίσουμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Αντωνίο Ταγιάννη. Ε, Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω στα γαλλικά όλου του βουλευτέ που υποστήριξαν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την προσήλωσή τη να ακούστουν η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή υπέρ της ελευθερίας στο διαδίκτυο. Όχι μόνο του συστήματος, αλλά και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Αντιπρόεδρος ε, Κρούς θα ενημερωθεί ε, για τη συζήτηση. Αλλά πρέπει να σας πω το σχέδιο ψηφίσματος που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έβλαπτε τις προσπάθειες που καταβάλει εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να τις δώσει το Συμβούλιο διαπραγματευτική εντολή στα πλαίσια της Διεθνούς Διάσκεψης WICIT. Σύμφωνα με το άρθρο 218 ε, της Συνθήκης Τονίζω, η Ευρώπη θα πρέπει να έχει στεναρή αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το ελεύθερο και χωρίς παρεμβάσει διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Πρόεδρε, το λόγο έχει του Συμβουλίου ο κύριος ε, Λουκάς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή έχω καταχραστεί λίγο το χρόνο στην αρχική μου τοποθέτηση, θα είμαι πολύ σύντομο. Δεδομένη τη σημασία των συνεδρίων όπω το WeKit, για το μέλλον του ψηφιακού θεματολογίου για την ευρώπη οι απόψει όλων των θεσμικών οργάνων είναι ευπρόσδεκτε. θα πρέπει επίση να έχουμε μια σαφή κατανόηση του τι θα πρέπει να είναι ο ρόλο αυτών των συνεδρίων με μια τέτοια ευρεία εκλογική περιφέρεια σαν ένα τομέα όπου η τεχνολογία και το περιεχόμενο εξελίσσονται τόσο γρήγορα δεν πρέπει να πάει σε μικρορύθμιση αλλά να διασφαλιστεί ότι οι αναθεωρημένοι κανονισμοί παραμένουν σε ψηλό επίπεδο στρατηγικά και τεχνολογικά ουδέτεροι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε για το WICIT και για την πρόθεσή σας για έγκριση του σχετικού ψηφίσματος. Κλείνοντας, να επαναλαμβάνω ότι η Προεδρία έχει δεσμευτεί πλήρως να διευκολύνει την εκπροσώπηση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντουμπάι η οποία θα ευθυγραμμίζεται με το κεκτημένο και θα υποστηρίζει μια πιο δυναμική ψηφιακή Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Έλαβα τρεις προτάσεις ψηφίσματος για την παράταση αυτή της συζήτηση. Η συζήτηση κηρύσσεται περιομένη, ε, περιομένη. Η ψηφοφορία θα διεξαρθεί την 5η 22 Νοεμβρίου. Οι συνεδρίες διακόπτεται ως την 21η ως 9 η ώρα. Καληνύχτα.